Colleagues, I kindly ask you to take your seats now. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι. Ε, καθυστέρησαμε γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε και κλεισμένα των θυρών. Και τώρα θα δείξουμε το ίδιο ενδιαφέρον, με ναι, πριν, για το επόμενο σημείο, που είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση στη Σομαλία και την κατάσταση ασφάλειας στη Σομαλία. Και καλωσορίζω τον συνταγματάρχη Χωακίν Μπέρνς, που είναι τμήματάρχης ενός ε, μεγάλου ονόματος, επιχειρήσεις ε, για το σχεδιασμό απόκρισης της κρίσης και τις τρέχουσες επιχειρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, είναι χαρά και τιμή να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την ε, αποστολή κατάρτισης στη Σομαλία. Είναι μία από τις τρεις που έχουμε. Ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τρεις ε, αποστολές στην Αφρική στρατιωτικού τύπου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για αυτό το θέμα μετά από το προηγούμενο τόσο ενδιαφέρον θέμα με το τόσο καλούς ομιλητές. Θα κάνω ό,τι μπορώ ούτω ώστε να σας τραβήξω την προσοχή που, για αυτό το θέμα που επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πριν ξεκινήσω όμως, θα ήθελα να σας πω ποιος είμαι. Είμαι ο Προύνς, ε, είμαι παντρεμένος, τρία παιδιά έχω. 14 ε, μετακομίσεις κάναμε στη στρατιωτική μου καριέρα με την οικογένεια. Να μην τα εξηγήσω όλα αυτά. Ε, κάποια αναφέρονται. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι στις Βρυξέλλες. Χαίρομαι και εγώ και η οικογένειά μου. Εξήγησε η πρόεδρος ε, τη θέση μου στην αποστολή αυτή, αλλά παράλληλα δουλεύω για το στρατιωτικό σχεδιασμό ε, για ένα τμήμα που δημιουργήθηκε πέρσι τον Ιούνιο. Είμαι υπεύθυνο ε, στα πλαίσια αυτού του Ινστιτούτου μου για, και για τις τρεις αυτές αποστολές. Έρχομαι εδώ υπό τη διπλή μου ιδιότητα. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Θα σας κάνω μια Σύντομη ενημέρωση για την πολιτική κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κατάσταση στη χώρα είναι πάρα πολύ ευάλωτη, δύσκολη, αλλάζει γρήγορα. Έχουμε τα ομόσπονδα ε, κρατήδια με βάση τις φυλές. Έχουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που προσπαθεί να δημιουργήσει ομοσπονδιακούς θεσμούς και οργάνωση που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν αντιστάσεις από αυτές τις ε, περιφερειακές ε, από τους περιφερειακούς αυτούς φορείς. Αυτό είναι ένα συνεχές πρόβλημα και έχουμε επίσης και ένα πολύ σημαντικό θέμα της μετάβασης από την αμνηστία σε μια κατάσταση που να υπάρχει ασφάλεια. Έχουμε την Άρμισον που είναι διάφορες δυνάμεις, ε, μαχητικές δυνάμεις από πέντε αφρικανικές χώρες για να εξασφαλίσουν ασφάλεια στην περιοχή, για να καταπολεμηθούν οι τρομοκρατικές ε, ομάδες. Ε, έχουμε το Αλσαμπά που είναι πρόσκειται στην Αλκάιντα. Θα πρέπει με τους άλλους διεθνείς φορείς να εξασφαλίσουμε ότι η Σομαλία έχει δικέ τη δυνάμει ασφαλεία στο μέλλον, ούτω ώστε να ασχοληθεί με την εθνική τη ασφάλεια και να μην βασίζεται στην υποστήριξη που θα τη δίνουν άλλοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο πληρώνουμε 240 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ε, στρατιωτικών δυνάμεων στη Σομαλία. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά μας αυτή για την ασφάλεια της χώρας. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη όπου αυτό το σχέδιο μετάβασης θα συζητηθεί εκ νέου και η διάσκεψη ψηλού επίπεδου θα, σε αυτή θα συμμετάσχει ο κύριος Σαβάνο που είναι ε, το νούμερο 2 της ε, υπηρεσίας μου, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, καθώς και ο Πρωθυπουργό της Ομαλίας ο οποίο είναι και υπεύθυνο για αυτό το σχέδιο μετάβαση για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Πάμε στην δική μας αποστολή κατάρτισης, που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, το 2011, στην Ουγκάντα, θα θυμάστε ίσω, και συνεχεία πέρασε στο Μογκαντήσου το 2013-2014. Είναι μια αποστολή συμβουλών, παροχή συμβουλών και κατάρτισης. Εδώ βλέπετε τα καθήκοντά μας, που είναι να δώσουμε πολιτικές και στρατηγικές ε, στρατιωτικές συμβουλές που σημαίνει ότι η σύμβουλή μας είναι σε θέσεις κλειδιά ή τουλάχιστον πλαισιώνουν ε, τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά ε, στο Υπουργείο Άμυνας και στις, ε, στο στρατό της Σομαλίας για να τους δίνουν σημαντικές συμβουλές. Προπολογισμό, θέματα προσωπικού, επιχειρησιακά θέματα. Τους συμβουλεύουμε τους δίνουμε συστάσεις και παράλληλα κάνουμε και κατάρτιση ε, μονάδων, εκπαίδευση και κατάρτιση μονάδων που μας υποδεικνύουν αρχές. Τους δίνουμε εκπαίδευση ούτω ώστε, μιλάμε για ομάδες ε, πεζικού, και αυτή τη στιγμή έχουμε εκπαιδεύσει τρεις λόγους ε, πεζικού, που μοιάζει να είναι λίγο, όμως είναι μονάδες, είναι λόχοι που αποτελούνται από διάφορες φυλές. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατιώτε από όλε τι περιοχέ τη χώρα, από όλε τι φυλέ για να δημιουργήσει ένα πραγματικό σομαλικό στρατό, για να αισθάνονται ότι είναι ο πραγματικό στρατός της ε, μελλοντική σομαλική κυβέρνηση. Καλύτερα λίγου και καλού, λίγου και παραγωγικού, αλλά πολλού και ανεξέλεγκτου. Ένα από τους λόγου, ε, καταπολεμάει το Al-Shabaab αυτή τη στιγμή. Ο, ο άλλος λόγος χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο ω φρουρά. Καλό θα είναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση αυτοί οι στρατιώτες, αφού τους χρησιμοποιεί για την προσωπική του φρουρά. Και επίσης ε, εκπαιδεύουμε και μια άλλη μονάδα που θα τη χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Πήραμε εντολές από τον Σομαλικό στρατό ε, πρόσφατα να εκπαιδεύσει και άλλες δυνάμεις. Όσον αφορά το συμβουλευτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων μας, είμαστε πολύ δραστηροί. Προσπαθούμε λοιπόν να τους δώσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες ποια, α, ποιος είναι ο ρόλος που παίζουμε. Αφορά το Υπουργείο Άμυνας, ούτως ώστε να υπάρχει μια γενικός έλεγχος ε, πολιτικός στατιωτικός που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και μετά πάμε και επίτοπου για θέματα οργάνωσης επιμελητίας. Πώς να δώσουμε υποστήριξη σε μονάδες που είναι ανεπτυγμένες επί τόπου. Να είμαστε σίγουροι ότι πληρώνονται και δεν θα πάνε στην άλλη πλευρά λόγω ε, ελήψεως ε, χρημάτων, ελήψεως μισθών. Όλα σχετίζονται με αυτές τις στατιωτικές πτυχές και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό παρέχουμε εκπαίδευση για τους μελλοντικούς εκπαιδευτές των Σαμαντών. Να εκπαιδεύεις τον εκπαιδευτή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε την πρόθεση στο τέλος οι Σομαλοί να μπορούν να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τις μονάδες τους από τις διάφορες φυλές και από τα μόσπονδα κρατήδια ώστε να έχουν τελικά μια βιώσιμη δομή για αυτές τις δυνάμεις. Τώρα τα προβλήματα, οι προκλήσεις, ίσως ε, ήδη θα έχετε μάθει, θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαγνώσει ότι οι πολιτικές εντάσεις ακόμα είναι μεγάλο πρόβλημα για όλους στη χώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εφαρμογή ε, και υλοποίηση της μετάβασης όσον αφορά τις ομαλικές αρχές προς μια κατάσταση ασφαλή. Υπάρχουν πολλοί διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους και να τονίσω ότι έχουμε άριστες σχέσεις με τους Αμερικανούς επιτόπου έχουν μια ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Νέα πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ε, πέρσι το Μάιο στη διάσκεψη του Λονδίνου για την ασφάλεια και σε διάφορους τομείς προχωρούν οι Αμερικανοί και η δική μας εκπαιδευτική αποστολή είναι επιφορτισμένη με έναν από του κρίσιμου τομείς, δηλαδή να παράσχουμε υποστήριξη και συμβουλές ε, στο στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων της Σομαλίας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα μεταξύ άλλων και είναι ένα καλό σημάδι διεθνού συνεργασία. Αλλά πρέπει να αισθανθούν οι, το, οι ντόπιοι την ιδιοκτησία τους όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει δυστυχώς να πω ότι βασιζόμαστε στην υποστήριξη των κρατών μελών για να παράσχουμε τους αναγκαίους πόρους. Δηλαδή προσωπικό, ειδικό προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, για την ώρα αυτό μας απασχολεί ε, και στο στρατιωτικό σχεδιασμό. Χρειαζόμαστε περισσότερους συμβούλους, εκπαιδευτές και προσωπικό. Ε, μια στατηγική επισκόπηση συζητήθηκε αυτό σε πολιτικό επίπεδο ως ιδέα. Κοινή λογική είναι να συνεχίσουμε με την εντολή που μας ανατέθηκε για την εκπαίδευση για την επόμενη διετία μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 μαζί με την αποστολή μας στον πολιτικό τομέα και την επιχείρηση Αταλάντα που υλοποιείται σε αυτή την περιοχή και μπορώ να σας δείξω και κάποιες εικόνες πριν ολοκληρώσω, να δείτε πώς ε, μαζί κάνουμε την εκπαίδευση. Μ' αρέσει η φωτογραφία στα δεξιά, πάνω δεξιά, όπου δίνουμε αρβίλες, διότι συνήθως έρχονται με σαγιονάρες. Τους δίνουμε αρβίλες, τις επόμενες ημέρες ίσως δυστυχώς μετά από μέρες δεν επιστεύουν τις μπότες, τις χάνουν, χάνουν τις αρβίλες ε, και πρέπει να τους δώσουμε άλλες Μ' αρέσει αυτός ο τύπος εδώ, που ίσως είναι η πρώτη φορά που είδε αρβίλες. Είναι σημαντικό, αφορά την αξιοπιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιούμεθα μαζί με τους άλλους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου και αξίζουν οι προσπάθειες αυτές που καταβάλουμε για την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την βιωσιμότητα της χώρας ε, στο μέλλον. Εδώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Συνταγματάρχα για αυτή την εισαγωγή, την παρουσίαση που κάνατε και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ξεκινάμε τους συντονιστές και από τον κύριο Γκάλερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της εκπαιδευτικής αποστολής. Είδα και την ετήσια έκθεση για τις επιχειρήσεις στη Σομαλία. Πολιτικά νομίζω η Αφρικανική Ένωση με την αποστολή, την αμισόν ζήτησε πρώτα απ' όλα μια χρηματοδοτική στήριξη αναφέρατε τα 240 εκατομμύρια ευρώ το ερώτημα είναι βεβαίως τι θα γινόταν αν δεν το κάναμε εμεί, πιθανώ δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση από την ε, Αφρικανική Ένωση και το έφτραυστο κράτος ε, της Σομαλίας μάλλον ε, θα κατέρεε πάλι και θα είχαμε μόνο τις διάφορες φάρες που θα έλεγχαν μέρος της επικράτειας. Οπότε πρέπει να ενισχυθεί η Σομαλία ως κράτος όσον αφορά ναι. και την δική μας τη χρηματοδότηση και μετά βεβαίως πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η αποστολή αυτή ε, ανταποκρίνεται στην πολιτική βούληση της ε, κυβέρνησης. Και εκεί πέρα πραγματικά το ερώτημα είναι το εξής. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε στέκει είναι βιώσιμο. Οι Ολλανδοί νομίζω έχουν ήδη αποσυρθεί και σιγά σιγά θα αποσυρθούν και οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί είπαν ε, ότι υπάρχει περιορισμένη στρατιωτική αποτελεσματικότητα της αποστολής και στη γερμανική ανακοίνωση λένε ότι παρά τις ε, προσπάθειες ε, ο Σωμαλικός στρατός ε, αναπτύσσεται πάρα πολύ αργά και υπάρχουν ελλειπείς δομές. Αναφέρατε λοιπόν προβλήματα και στο νέο έργο, το CBSD, το Capacity Building for Security Development, ότι τουλάχιστον το μη στρατιωτικό κομμάτι θα, θα έπρεπε να προσεχτεί. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν εκεί ακριβώς Και βεβαίως αναρωτιέμαι όταν μιλάμε για τον προγραμματισμό του 2019 και 2020 με ποιον το προγραμματίζετε. Δεν ξέρω αν έχει νόημα δηλαδή να μιλάμε για διάθεση προσωπικού. Σας ευχαριστώ κύριο Βανόρντεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. όπως και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ντανζόν και ο κύριος Πάσκου, επισκεφθήκαμε την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη Σομαλία όταν ήταν στην Ουγκάντα, εδώ και κάποια χρόνια. Συνεχίζεται λοιπόν η αποστολή. Διρωτώ με ποιο είναι το νόημα. Φαίνεται ότι είναι μία από τις αποστολές εκείνες που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι κάτι κάνει. Καλό αυτό. Για την εικόνα. Αλλά τι πετυχαίνει από πλευρά στατιωτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι στατιώτες εκπαιδεύονται από την αποστολή και πόσο διαρκούν, πόσο μαθαίνουν τελικά, ενστερνίζονται τις γνώσεις αυτοί που εκπαιδεύονται. Ίσως δεν είναι θεμητό, θέτω το ερώτημα σε εσά. Ποιο θα ήταν ο αποφασιστικό αντίκτυπο για την κατάσταση της τι θα έπρεπε να κάνουμε. Η διεθνή κοινότητα είναι κάπως στο περιθώριο. Έχουμε παγωμένη σύραξη εκεί. Δηλαδή δεν αλλάζει η κατάσταση ασφαλείας στη Σομαλία. Φαίνεται να το έχουμε αποδεχθεί και είναι ατέρμονη αυτή η κατάσταση. Τι θα κάνουμε για να σταματήσει. Η απάντηση βέβαια σε αυτό θα ήταν κάτι δύσκολο, αιματηρό κλπ. να είναι κάτι πιο δραστήριο, πιο δραστικό. Πρέπει να συμβεί, αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν την πολιτική βούληση να πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Λούζινγκ έχει το λόγο. Ähm, Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα ακούστηκαν ήδη. Αναφέρατε ακριβώς ε, το θέμα αυτό του ότι ξεπερνάει η αποστολή τα όρια της. Τα είδα και στο ίντερνετ. Εκεί πέρα μιλάμε για 5.500 Σομαλούς ε, στρατιώτες που έχουν εκπαιδευτεί. Ε, πόσοι από αυτούς είναι στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Ποιος είναι ο αριθμός. Και είναι γνωστό πόσοι ε, στρατιώτες μετά πήγαν ε, στις διάφορες ένοπλες ομάδες ατάκτων. Αν μπορείτε να κάνετε κάποια εκτίμηση. Μετά υπάρχει η συνεργασία με τους Αμερικανούς που αναφέρατε. Διάβασα πριν από λίγες ημέρες πως η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε την έκθεση που λέγεται Deadly Assistance για την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε χτυπήματα με μη πανδρομένα αεροσκάφη. Όπου μιλάμε για την παροχή δεδομένων αναγνώρισης ε, σε στόχους στην Σομαλία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς ε, έχει ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ της αποστολής σας ε, και των δυνάμεων των ΙΠΑ και αν ανταλλάσσονται και δεδομένα που χρησιμοποιούνται μετά για χτυπήματα με μη επανδρομένα. Και τέλος αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γκάλερ το θέμα της αποτελεσματικότητας η κατάσταση ασφαλείας τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί, έχει βελτιωθεί, έχει παραμείνει σταθερή και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας εκτίμηση. Ο κύριος Γκάλερ ανέφερε ε, το ότι η Ολλανδία εγκατέλειψε την αποστολή για ποιο λόγο εκτιμάτε εσείς. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Έχει το λόγο. Ο κύριος Κάρβερ. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πάμε σε αυτά που είπε ο Γκάλερ. Για κάποιον που αντιλαμβάνεται τι γίνεται στη Σομαλία. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα όσον αφορά να λάβουμε υπόψη τη δομή που είναι βάση των φυλών στη Σομαλία και φαίνεται να έχει καταρρεύσει το σύστημα και οδήγησε σε αναρχία. Ερώτηση. Έχουμε μια προθεσμία. Δύο χρόνια περιθώριο. Και έχουμε επιθέσεις στο, της Σάσαμπαπ, στο Τζιμπουτί και στην Κένια. Τα δύο χρόνια μπορεί, αρκούν. Εάν η αποστολή που έχει δρομολογηθεί δεν καταλήξει εκεί που πρέπει, θα παραταθεί. Ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες. Thank Ευχαριστώ, κύριε Ντανζόν. Ευχαριστώ. Δυστυχώς, για μια φορά, πιστεύω, ότι ο τόνος που θα προσθέσω στη συζήτηση δεν θα είναι υποστηρικτικός σε μία από τις αποστολές μας ΚΕΠΑ. Ε, και εγώ θα ε, επικρίνω κάπως την όλη κατάσταση από συνάδελφος Βαν Όρντεν. Όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια παρουσία στο κέρας της Αφρικής και πιο συγκεκριμένα στη Σομαλία. Διερωτώ με για τις λεπτομέρειε της αποστολής και αυτή η αποστολή της εκπαιδεύσεως, η UTM, φαίνεται αποστολή άλλου τύπου την αποκαλώ. Έχουμε τη σημαία μας, εκεί κάτι κάνουμε, αυτό δίνει αποτελέσματα από τη θέμενη αξία. Ξέρω εγώ. Είναι αποφασιστική σημασία, σίγουρα όχι. Τι με συγκλονίζει λίγο. Ε, 8 χρόνια διαρκεί αυτή η αποστολή. Αυτή η διαδικασία κρατάει πάνω από δεκαετία. Θυμάμαι ότι πήγα στο Τζιμπουτί το 2008 όπου οι Γάλλοι ήδη εκπαίδευαν τους Σομαλούς στατιώτες. Η UTM ήταν ως επεκτάσεως ευρωπαϊκής του λόγω προγράμματος. Και εδώ και 10 χρόνια κάνουμε το πρόγραμμα αυτό και πάντα υπάρχουν τα ίδια ερωτηματικά. Να εκπαιδεύσουμε, θέλουμε τους εκπαιδευτές, να υπάρχει καλύτερη πλαισίωση, επίπεδο αξιοπιστίας, πώς εξακριβώνουμε ότι οι στατιώτες που εκπαιδεύσαμε μπαίνουν στον τακτικό σομαλικό στρατό και δεν μπαίνουν σε φιλετικά μορφώματα, μην μπουμε αλσαμπάμπ. Δεν ξέρω τι πρόοδο επιτυγχάνεται εκεί. Τα ίδια ερωτήματα υπάρχουν, ελάχιστε απαντήσει. Μας λέτε θα γίνει στατηγική αναθεώρηση. Αυτή η αναθεώρηση ακολουθεί άλλη αναθεώρηση. Και ξέρουμε εκ των προτέρων τα αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η χρηματοδότηση τη Αμισόμ είναι κάτι σημαντικό. Και αν δεν είχαμε χρηματοδοτήσει την Αμισόμ, σίγουρα η Αμισόμ θα κατέρε και η κατάσταση στη Σομαλία θα ήταν ακόμα χειρότερη. Και το UTM είναι κάτι αμφισβητήσιμο υποστήριξη της ε, επιχειρήσεως αυτής. Αν θέλουμε να ε, έχουμε αποτέλεσμα στο UTM κατανοώ τους πολιτικούς. στα κράτη-μέλη λένε ότι δεν θα στείλουμε προσωπικό σε αυτή την αποστολή, σε αυτή την επιχείρηση. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις τους. Δεν βλέπω πλέον ξεκάθαρα σε τι εξυπηρετεί αυτή η αποστολή. Ποια η σχέση μας με τους άλλους διεθνείς φορείς, που είναι πάρα πολλοί. Το κακόμοιρο το αεροδρόμιο του Μογκαντήσιο έχει πλημμυρίσει, έχει κατακλειστεί από τη διεθνή παρουσία. Μιλήσατε, κάποια πως Μιλήσατε για το στρατηγικό συμβούλιο του Υπουργείου Αμήνης της Σομαλίας. Λοιπόν, Έχουμε μία σύνοδο κορυφή, έχουμε διμερεί επαφέ, έχουμε του Βρετανού, του Αμερικανού που κάνουν πάρα πολλά, έχουμε του Τούρκου που κάνουν πάρα πολλά πράγματα για ακόμη περισσότερο από εμά εκεί. Έχουμε τι χώρε του κόλπου. Δεν το συζητήσαμε. Πρόσφατα το πρόβλημα μεταξύ Κατάρα, Σαουδική Αραβία και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε συνέπειε πάρα πολύ μεγάλε για τη Σομαλία που επέλεξε στρατόπεδο. Και να σταματήσουν κάποια προγράμματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ήταν μεγάλος προμηθευτής βοηθείας και ενισχύσεως και συμβουλών σε στρατιωτικό επίπεδο. Ποια η διάδρασή μας με τους άλλους ε, διεθνείς φορείς. Βλέπουμε το βάρος των άλλων φορέων και πολύ συχνά είναι πολύ παλιοί όσον αφορά τις δομές της Ομαλίας. Και πώς συγκρίνεται αυτό με τη δική μας ε, παρουσία μέσω της UTM. Ίσως είναι μηδαμινή αυτή η παρουσία μας εκεί. Ήταν η τελευταία παρέμβαση Ευρωβουλευτών, λέει η Πρόεδρος. Ε, στα, ε, συνταγματάρχα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες και σημαντικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα από την στρατιωτική σκοπιά, γιατί αυτό μπορώ εγώ να πω. Τα πολιτικά ερωτήματα βεβαίως είναι δικά σας ε, ζητήματα και αρμοδιότητα ειδικά όσον αφορά και την δημιουργία της ε, δύναμης που είναι σημαντική πτυχή. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τα κράτη μέλη να δώσουν τις δυνάμεις που έχουν αποφασίσει. Ωραία, λοιπόν. Τώρα όσον αφορά την οικονομική στήριξη στην Άμισομ, ναι, ετέθη το ζήτημα. Ε, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 240 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Θα μειωθούν και άλλο αναλόγως με την επιτυχία, αλλά χωρίς αυτήν την στήριξη είμαι πεπισμένος πως οι χώρες ε, που συνεισφέρουν ε, δεν θα θέλουν τόσο. Ίσως οι γειτονικέ χώρες να ενδιαφέρονται περισσότερο για να παρέχουν και για να εξασφαλίζουν και κάποια οικονομική επιρροή αλλά και για να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Αλλά χωρίς οικονομική στήριξη της Ένωσης ε, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Η μετάβαση της Άμισομ είναι, το ανέφερε, είναι ένα θέμα κλειδί. Δύο χρόνια τώρα είναι μια κατευθυντήρια γραμμή αν θέλετε. Όλοι οι διεθνείς ε, φορείς ε, συμφωνούν ότι θα πρέπει η μετάβαση να γίνει με βάση κάποιους όρους. Δηλαδή μόνο αν ο Εθνικός Στρατός Σομαλίας και οι δυνάμεις ασφαλείας ε, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ευθύνες, τότε θα αποσυρθεί η Άμισομ από τις σχετικές περιοχές. με βάση κάποιους όρους. Λοιπόν, τώρα είμαστε μαζί με την αντιπροσωπεία. Και βεβαίως ε, προσπαθούμε ακριβώς να βρούμε το μίσο που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να βρούμε το μίσο για να αναλάβουν την ευθύνη οι Σομαλοί. Όχι μόνο ο στρατός, αλλά και την διοίκηση γενικότερα. Οπότε είμαστε με μια αποστολή εκπαίδευσης και βεβαίως για να στηρίξουμε ακριβώς την παροχή ασφαλείας. Λοιπόν, με την απόσυρση τώρα της Ολλανδίας και της Γερμανίας, το καλύτερο είναι να ρωτήσετε τις χώρες. Είμαι ο εξωματικό βεβαίω, τα ξέρω αυτά, αλλά εδώ έχω έρθει ω Ευρωπαίο. Έχω τελείω διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι αν συγκρίνουμε την κατάσταση ασφαλεία, Όπω να αναφέρατε, με την κατάσταση πριν από 5 ή 10 χρόνια, όπου μιλούσαμε για ένα διαλυμένο κράτο, αποτυχημένο κράτο. Ε, που αποτελούσε καταφύγιο τρομοκρατών, έχει αλλάξει, εντάξει, ίσως όχι αρκετά γρήγορα, αλλά αλλάζει. Και υπάρχει πρόοδος. Επίσης αναφέρατε κάποια πρόοδο, αλλά δεν είναι αποφασιστική. Ε, είναι μακροπρόθεσμο το θέμα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξαντληθεί σε 3-5 χρόνια, αλλά σε 10-20 θα έλεγα. Ναι. Τώρα, ε, στα άλλα ζητήματα, τα πολιτικά. Πράγματι έχουμε βρει κάποια έργα, δημιουργούμε υποδομές, ε, φτιάχνουμε γραφεία και διοικητήρια, επίσης μέσα επικοινωνίας, μαζί με την Κομισιόν, ε, με μια κοινή προσέγγιση, στρατιωτική και πολιτική πτυχή έτσι ώστε το κράτος Σομαλίας να αποκτήσει κάποιες δυνατότητες ελέγχου. Κάτι λοιπόν υπάρχει εκεί. Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα, αλλά από τη δικιά μας τη σκοπιά τη στρατιωτική θα έλεγα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για οικονομική στήριξη από την Κομισιόν που μπορεί οπωσδήποτε να αναπτυχθεί περισσότερο στο μέλλον. Αλλά έχει ξεκινήσει και βλέπουμε κάποια πρόοδο. Τα επιτεύγματα. το θέμα των 5.000 εκπαιδευμένων ε, στρατιωτών. Ναι, νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρούμε πού βρίσκονται τώρα, τι κάνουν. Γιατί όταν τους εκπαιδεύσαμε στην ε, πρώτη φάση, στην Ουγκάντα μάλιστα, δεν υπήρχε κάποιος μηχανισμός ελέγχου για να δούμε το που πήγαιναν μετά και όπως είπα, το κλειδί είναι ότι αυτοί οι στρατιώτες ε, θα πρέπει να πληρώνονται και από το κράτος, ε, να προσληφθούν δηλαδή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να θέσετε στις αρχές της χώρας. Δεν μπορώ λοιπόν ούτε να μαντέψω ούτε εικασίες να κάνω. Αν έχουμε τώρα επηρεάσει αποφασιστικά την σύγκρουση, ε, θεωρώ ότι υπάρχει πρόοδος σε σχέση με τα όσα είχαμε πριν από 10 χρόνια. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση για ένα ομοσπονδιακό κράτος ή κάτι τέτοιο. Πριν από 5-10 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο οι φάρες ε, και τρομοκρατία. Οπότε κάτι βλέπω και μπορούμε βεβαίως να εκπαιδεύσουμε τις ομάδες αυτές. Έχουμε εκπαιδεύσει ήδη τρεις ε, λόχους ε, από, που είναι στελεχωμένοι από όλες τις φάρες και είναι επιχειρησιακοί. Θεωρώ λοιπόν ότι Έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, ίσως όχι όσα περιμέναμε, αλλά χρειάζεται μια πιο μακροπρόθεσμη, θα έλεγα, προσέγγιση στη χώρα αυτή. Για να τα υπόλοιπα, διεθνής ε, συνεργασία. Όπως ανέφερα, οι Αμερικανοί είναι πολύ ενεργοί σε μια συνολική προσέγγιση ασφάλειας ε, και συνεργασίας και βεβαίως ασκούν και πίεση στην ε, κυβέρνηση της χώρας που απαιτείται και εμείς είμαστε μαζί τους ε, σε στενή επαφή, αναλαμβάνουμε ευθύνε σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είπα, παρέχουμε συμβουλές στο Γενικό Επιτελείο, Και υπάρχει και συνεργασία και με την Τουρκία που έχει παρουσία στη χώρα. Και συνεργάζεται μαζί μας και με την διεθνή κοινότητα και με μας. Για την ώρα είναι θετικό αυτό το μήνυμα. Τώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους Αμερικάνους, ε, η αποστολή μας ε, δεν ανταλλάσσει δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στόχους. Είμαστε μη εκτελεστική αποστολή. Δεν έχουμε δυνατότητες αναγνώρισης ε, και πληροφοριών μόνο για προστασία, αυτοπροστασία της δύναμής μας. Δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή πληροφοριών ε, όσον αφορά την στόχευση μη επανδρομένων ε, αεροσκαφών. Λοιπόν, η επόμενη εντολή που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο θα εστιάσει περισσότερο σε μια αύξηση των δυνατοτήτων και στην εκπαίδευση για να μπορούν να εκπαιδεύουν όπως εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά με δικούς τους εκπαιδευτές. Και έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο Μογκαντίσου ήδη με 20 συμμετέχοντες και κάποιοι από αυτούς μένουν στον χώρο της εκπαίδευσης και εκπαιδεύουν τις επόμενες μονάδες και εμείς μπορούμε ακριβώς εκεί να τους συμβουλεύσουμε στα της εκπαίδευσης. Είναι μια σταδιακή διαδικασία. Εγώ βλέπω κάποια πρόοδο. Είμαι πεπισμένο ότι είναι σωστή η διαδικασία, αλλά συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και σας ε, καλό να σκεφτείτε όταν ε, αποφασίζουμε μια τέτοια αποστολή να παρέχουν τα κράτη-μέλη τους απαραίτητους πόρους. Ελπίζω λοιπόν να απάντησα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε συνταγματάρχα. Λοιπόν, Ας χειροκροτήσουμε τον ομιλητή μας, παρακαλώ. Thank you and thank you for this point of Σας ευχαριστώ. Καλύφθησαμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μας απομένουν αρκετά ακόμα για σήμερα στην πρωινή συνεδρίαση αλλά και στην απογευματινή συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να παραμείνετε. rather. They're all here. This is Mr. Stirnon, the chair of the committee, Mrs. Fatigue. I'm sorry. sorry. Hello. Colleagues, please be seated. Before we... Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Πριν πάμε στο επόμενο σημείο για την εξαγωγή όπλων. Να σας ενημερώσω συντομία όσον αφορά την αποστολή μας στην Βοσνία Ριζεγοβίνη. Η αποστολή της Επιτροπής μας πραγματοποιήθηκε από τις 3 μέχρι 5 Απριλίου φέτος. Εκτός από την υποφαινομένη υπήρχαν και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών ομάδων, ΕΛΚ, ο κ. Κρίστιαν Νταν Πρέντα, S&D, τον Ίνο Πίτσουλα και η κυρία Βαλέρο, συντονίστρια των Πρασίνων. Λυσμόνησα κάποιον. Όχι, όχι. Κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο ημερών, διότι φτάσαμε αργά το απόγευμα, στις 3 του μηνός, μπορέσαμε να ενημερωθούμε πλήρως από την ε, αντιπροσωπεία μας εκεί. Βασικός στόχος ήταν να αναλύσουμε τις ε, επιχειρήσεις της U4 Αλθεία που ε, βρίσκεται εκεί. και των διοικητών του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε την ενημέρωση. Το πολιτικό πρόγραμμα ξεκίνησε με συνάντηση υψηλού επίπεδου με τον πρόεδρο της προεδρ... τον κύριο Ζερμπέγκοβιτς, τον πρόεδρο της Βοσνίας και συναντήσαμε και εκπροσώπους ε, άλλων μελών ε, της κυβερνήσεως Κατά τη διάρκεια της αποστολής μπορέσαμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης αντιπροσωπεία της κοινωνίας των πολιτών επίσης και επιχειρηματίες, επιχειρήσεις μάλλον, που εταιρείε που ασχολούνται με την αποναρκοθέτηση και έγινε μια παρουσίαση της αποναρκοθέτησης ε, έγινε μια επίδειξη πλευρά των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης όσον αφορά την αναφέρουση των αρκών επισκεφθήκαμε το αρχηγείο της U4 και το αρχηγείο του στρατού της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, ε, έξω από το Σεράγεβο. Γενικά, αυτά κάναμε κατά διάρκεια του τριημέρου. Συναντήσαμε επίσης, ως ήθιστε, το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διαπιστευμένα μέλη διπλωματικού μας σώματος που ε, βρίσκονται στο Σεράγεβο και σε μια ξεχωριστή συνάντηση είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Αμερικανό πρεσβευτή και τον Ελβετό πρεσβευτή ήταν πληρέστατη η τροφοδότησή μας σε πληροφορία και θα ενημερωθείτε διόντως, θα ετοιμαστεί μια σχετική έκθεση. Σύντομα θα σας δώσουμε μια έκθεση των πεπραγμένων στην αποστολή αυτή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσουμε. Α, δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις. Κλείσαμε, ολοκληρώσαμε αυτό. Τελικά πρέπει να επανεξετάσουμε τα θέματα ασφαλείας των Δυτικών Βαλκανίων μπορέσαμε να επισκεφθούμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη σε μια δυσχερέστατη περίοδο χρονική που προηγείται των γενικών εκλογών. Η πολιτική κατάσταση όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιόδους ήταν πολύ τεταμένη. Όλοι μας εκφράσαμε μεγάλη ανησυχία. Φυσικά συναντηθήκαμε με σημαντικούς ε, συνομιλητές του Κοινοβουλίου και μάλιστα και των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου και τη Γερουσία και την ε, Βουλή της Βοσνίας ε, της Βουλής της Βορσίας Ζεγοβίνης και συναντηθήκαμε με μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών, ειδικά την Επιτροπή ε, Αμυντικών Υποθέσεων. Μπορώ λοιπόν εδώ να κλείσω αυτή τη σύντομη ενημέρωση και να πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση με πανελίστες για τις παγκόσμιες τάσεις ε, στις εξαγωγές όπλων. Ένας ομιλητής δεν έχει έρθει ακόμα. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρέμβασή του στο τέλος. Μιλάμε για την κυρία Καρολάιν Κλίφ, που είναι πρόεδρος της ΚΟΑΡΜ και της ΣΕΚΠΟΛ. Θα έρθει αργότερα. Έχουμε δύο ακόμα μιλητές. Έναν από τη Βαρκελόνη, τον κύριο Μαρία Βιέγιας Αρινιού, Αρινιού που εκπροσωπεί το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, μια σχολή που ασχολείται με την έρευνα για την ειρήνη και τον κύριο ζορδί Κάλβο Ρουφάγγες. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομα. που εκπροσωπεί το κέντρο ΔΕΛΑ της Βαρκελόνης. Είναι ερευνητή και συντονιστής. Ο κύριος Αρίνιο είναι ερευνητής στη σχολή στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και ο κύριος Χριστόφ Στιερνού από την ομάδα GRIP, από το κέντρο GRIP. Πολύ ωραία, θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις τους. Α, ήρθε και η κυρία Καρολάιν Κλίφ, πρόεδρος της COARM, που εκπροσωπεί τη ΕΚΠΟΛ εντός της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Κλειφ. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στη Μέση αλλά και τα προηγούμενα ήταν πολύ σημαντικά και είχαμε μακροσκελή συζητήσεις. Κυρία Κλειφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ και όλους τους ε, καλεσμένους. Ναι, κυρία Πρόεδρε, όπως, όπως εξήγησε και η κυρία Πρόεδρε, είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Ε, προεδρεύω στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εξαγωγή συμβατικών όπλων να εξηγήσω ότι σε αντίθεση με πολλές ε, άλλες ε, ομάδες εργασίας ε, δεν είμαστε γεωγραφική ομάδα, δηλαδή έχουμε προσώπους από τις πρωτεύουσες, συνεδριάζουμε μια φορά το μήνα πλην Αυγούστου, οπότε έχουμε γύρω στις 10 συνεδριάσεις το χρόνο. Να σας τα εξηγήσω δηλαδή αυτά γιατί 10 συνεδριάσεις το χρόνο δεν είναι και πάρα πολλές. Ε, τουλάχιστον. Έτσι θεωρώ εγώ που προεδρεύω. Να ξεκινήσω τις, εξεξηγώντας τις αρμοδιότητές μας αφορά την ε, στρατιωτική τεχνολογία, οπότε είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Από την άλλη, θα ξέρετε βεβαίως πως για τα αντικείμενα διπλής χρήσης η αρμοδιότητα είναι της Ένωσης, ε, συγκεκριμένα εδώ της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο που βρισκόμαστε όσον αφορά την κοινή θέση για την ε, εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας ε, η κοινή θέση 2008-944 να αναφερθώ λοιπόν το τι έχουμε κάνει και τι θα μας απασχολήσει το ερχόμενο έτος. Πρώτα απ' όλα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης στηρίζουμε ιδιαίτερο στην συζήτηση τέτοιων ζητημάτων με τους ενδιαφερομένους. Αναγνωρίζουμε την σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και θεωρούμε βεβαίως ότι έχει μεγάλη σημασία ο δημοκρατικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Το πλαίσιο της κοινότητας περιστρέφεται γύρω από την κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε το 2008 θα επανέλθω σε ένα λεπτό στην προτεραιότητά μας που είναι βεβαίως η επαναξιολόγηση της κοινής θέσης. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο είναι μοναδικό, βασίζεται στην εθνική ευθύνη των κρατών μελών, στην αδειοδότηση, μαζί βεβαίως με την αξιολόγηση κινδύνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου που καθορίζονται είναι συνολικά, καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τον κίνδυνο παρεκτροπής των όπλων και την απειλή στην εσωτερική σταθερότητα. Από την πλευρά λοιπόν των εσωτερικών ευθυνών, ο κοινός μας στόχος είναι να υπάρξει μια σύγκληση των εθνικών πολιτικών εξαγωγών όπλων. Πώς στηρίζουμε λοιπόν αυτήν την σύγκληση στην πράξη. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, έχουμε μια, τα κοινά κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου. Η καθημερινή τους εφαρμογή στηρίζεται σε κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Ναι, ναι, βέβαια. Να μιλήσω πιο σιγά. Λοιπόν, τέσσερα στοιχεία. Τα στοιχεία, τα κοινά κριτήρια αξιολογήση κινδύνου, η καθημερινή του εφαρμογή από τους αρμόδιου που στηρίζεται σε κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ σε, κάποιες, σε έναν οδηγό περιέχονται που αναθεωρήθηκε το 2015 για να εφηγραμμιστούμε με την σχετική συνθήκη Δεύτερον, ε, κοινό ορισμός του τι θεωρούμε όπλα. Είναι ο κοινό στρατιωτικός κατάλογος που ενημερώνεται κάθε χρόνο και η τελευταία ενημέρωση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών στις 26 Φεβρουαρίου και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 15 Μαρτίου. Το τρίτο στοιχείο αφορά ακριβώς ε, τις πληροφορίες για την άρνηση. Όταν απορρίπτεται δηλαδή μια συναλλαγή από ένα κράτος μέλος, το κοινοποιεί στα άλλα κράτη-μέλη μαζί με τους λόγους. Κατόπιν ε, τα κράτη-μέλη το συνυπολογίζουν αυτό στην πολιτική εξαγωγών τους όταν εξετάζουν ε, παρόμοιες συναλλαγές. Αυτό έχει αναπτυχθεί στα μέσα του 2015 για να υπάρξει μια ξεχωριστή πλατφόρμα που θα λειτουργεί η υπηρεσία μας για να έχουμε ακριβώς αυτές τις πληροφορίες. Αυτό το δέχτηκαν θετικά τα κράτη-μέλη και η πλατφόρμα ενημερώνεται τακτικά και οι νέες προτάσεις ε, συζητούνται με τα κράτη-μέλη. Τέταρτον, έχουμε τις συνεδριάσεις ε, της αρμόδιας ομάδας εργασίας που αφορά ακριβώς εξαγωγές σε ευαίσθητους ε, προορισμούς Όσον αφορά την διαφάνεια, η κοινή θέση απαιτεί οι εξαγωγές να αναφέρονται ετησίως σε αυτήν η ετήσια μας έκθεση. Η 19η ετήσια έκθεση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου στην επίσημη εφημερίδα. Να σας πω ότι, γιατί γνωρίζω ότι Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ετήσια έκθεση ειδικά από την κοινωνία των πολιτών. Είναι διαθέσιμη όταν εγκριθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών γιατί ανεβαίνει στην σελίδα. Γνωρίζω όμως ότι πολλοί ε, την κοιτάνε μόνο όταν δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα αλλά ε, μπορεί να περάσει χρόνος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ε, φάσης. Με την έκθεση αυτή συνεισφέρουμε στην ε, διαφάνεια και διαδίδουμε δεδομένα για τις ε, περαιτέρω συζητήσει. Από την ευρύτερη διεθνή σκοπιά, το αρχείο αυτό διαφάνειας είναι, θα έλεγα, η εξαίρεση παγκοσμίω. Μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες και λίγες άλλες, όπως είπα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς, δημοσιεύουν δεδομένα για τις εξαγωγές όπλων και τα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι τα μόνα τα οποία δημοσιεύουν και τις απορρίψεις άδειας εξαγωγής. Βεβαίως, πάντα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει στο μέλλον, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα εξή. Πρώτα, από όλα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ιουλίου 2015, η Επιτροπή μας πρέπει να επαναξιολογήσει την εφαρμογή της κοινή θέση και την εκπλήρωση των στόχων της το 2018. 10 χρόνια δηλαδή μετά την έγκρισή της. Οπότε έχουμε ένα σοβαρό καθήκον για την ομάδα μας φέτος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ για περαιτέρω σύγκληση και συνεργασία στον τομέα του υλικού πολέμου. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να διορθώνονται τα λάθη και να προσθέτουμε νέες ε, λειτουργίες, παραδείγματος χάρη ένα μενού με το οποίο θα μπορούν να ανεβάζουν πληροφορίες ε, τα κράτη-μέλη, πληροφορίες οι οποίες κατά κανόνα δεν ε, παρέχονται σε άλλα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να φορούν κάποιον έμπορο όπλων, ο οποίος ανησυχεί κάποιο κράτος. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε την 20η ετήσια έκθεση, τα δεδομένα δηλαδή του 2017, για να δημοσιευτεί πριν το τέλος του 2018. Και πρέπει να διασφαλίσουμε την έγκαιρη έγκριση του ενημερωμένου καταλόγου. Να συνεχίσουμε επίσης να διαχειριζόμαστε τις ε, δραστηριότητες μας προς τα έξω, που είναι δύο. Η μία φορά τις χώρες της κοντινής γειτονίας μας και μετά έχουμε και εντατικές επαφές με χώρες που είναι συμβαλόμενα μέρη της συνθήκης εμπορίου όπλων. Μπορώ να σας πω περισσότερα αργότερα, όχι τώρα γιατί ε, όπως είπαμε ο χρόνος πιέζει. Πρέπει να φροντίσουμε οι νέες εξελίξεις, παραδείγματος χάρη έλεγχη μετά την αποστολή, έναχος μικρών όπλων κτλ. να ε, αντικατοπτρίζονται επαρκώς και να υπάρχει συνεργασία με τρίτες χώρες και βεβαίω ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, την βιομηχανία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, η κοινή θέση ξεκαθαρίζει ότι η αδειοδότηση είναι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει ή να αμφισβητήσει τέτοιες αποφάσεις, όμως η κοινή θέση στηρίζει την μεγαλύτερη σύγκληση με κάποια κοινά στοιχεία και διαμοιρασμό των πληροφοριών. Άρα η σύγκληση είναι κάτι το οποίο είναι διαρκώς ένα έργο εν εξελίξη. Με συγχωρείτε αγαπητή κυρία. Θεωρούμε ότι κάποια από τα βασικά επιτεύγματα της κοινής θέσης ε, είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια σε ζητήματα εξαγωγής όπλων. Οι συζητήσει μας ε, σήμερα, και σα ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε, δείχνουν ε, πώ οι πληροφορίε είναι διαθέσιμες στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξεταστούν. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη ευθύνη των αρμοδίων αρχών. Το, πλήγμα, το πλέγμα αυτό είναι η ουσία της ε, κοινή ε, θέσης στο υψηλότερο ε, επίπεδο της συνθήκης ελεγχόπλων. Σας ευχαριστώ. I'm sorry, I have to wait a minute. Ευχαριστώ. Το, το κουμπί, είναι... Okay, thank you. Thank you. Madam, I would like to thank you for this uh, very brief, concise and, and very clear. Ευχαριστώ κυρία μου για την πολύ σύντομη και πολύ σαφή δήλωση για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις δράσεις της. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Μαρία Βιγέγιας Αρίνιου από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, ε, ερευνητή. Έχει τον λόγο. Και ο άλλος. Α, όχι, όχι, έκανα λάθος. Δεύτερος θα μιλήσει ο κύριος Αρίνιας. Ο κύριος Ζορντί Κάλβο θα μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που δεχτήκατε τη συμμετοχή μας σε αυτό το φόρουμ και που μας επιτρέπετε να παρουσιάσουμε τις εκθέσεις που έχουμε ετοιμάσει ε, στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου ΠΑΟΥ, ε, του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της ε, Βαρκελόνης για τις εξαγωγές όπλων από την Ευρώπη σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Πρόκειται για εκθέσεις όπου συνδυάζουμε διάφορα στοιχεία για τις εξαγωγές όπλων ευρωπαϊκών όπλων με τα στοιχεία που έχουμε για, τα, για τις χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Συνδυάζουμε αυτά τα στοιχεία. Θα τα παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο οι δυο μας. Θα παρουσιάσω λοιπόν τα στοιχεία για τις εξαγωγές όπλων καταρχήν και ο Μαρία Βιγέγιας θα παρουσιάσει ε, στοιχεία για τη σειράξεις για την, τον προορισμό των όπλων αυτών από την Ευρώπη. Ο στόχο των εκθέσεων αυτό που θα σας παρουσιάσουμε είναι καταρχάς να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της κοινή θέση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Κλίφ και να εφαρμοστούν τα κριτήρια για την αδειοδότηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας εξαγωγής όπλων λαμβάνοντα υπόψη ακριβώς εκείνα τα κριτήρια. Πρέπει να βλέπουμε που υπάρχει αστάθεια, σύγκρουση, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάφοροι άλλοι κίνδυνοι που ανέφερε η κυρία Κλίφ. Η ανάλυση των εξαγωγών όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της επίσημης έκθεσης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένας κατάλογος επικαιροποιημένος με όλα τα υλικά που θεωρούνται, όλους τους εξοπλισμούς που θεωρούνται στρατιωτικοί εξοπλισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις αυτές που σας παρουσιάζουμε αναλύουν τις εξαγωγές όπλων το 2015, πολύ συγκεκριμένα. Και βλέπουμε και την εξέλιξη στον χρόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν ως, ε, με σημείο αφετηρία στη χρονιά 2003, γιατί από τότε έχουμε αρκετές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσει συγκρίσεις για τις τάσεις των ε, εξαγωγών ευρωπαϊκών όπλων. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, θα μιλήσω για τις εξαγωγές λοιπόν όπλων και έχω να σας πω καταρχήν ότι υπάρχει μια αύξηση πολύ μεγάλη, εκρηκτική των εξαγωγών όπλων από το 2012, όπου τότε πολύ έντονα ε, αρχίσαμε δηλαδή να εκφράζουμε την πολιτική βούληση μέσω των αδειών έτσι, που δίνουμε στις εξαγωγές όπλων. Ε, η ίδια η βιομηχανία όπλων μας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιζητούσε αυτές τις άδειες για να εξάγει τα όπλα της ανά τον κόσμο. Υπάρχουν φυσικά κάποιες ελλείψεις στις εκθέσεις, γιατί δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίες από κάποια κράτη, δεν ξέρουμε τι άδειε έχουν δώσει σε κάποιους εξοπλισμούς. Και το 2015 λοιπόν βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν συμβάσεις για εξοπλισμούς, κυρίως στις κατηγορίες 2, 4, 9, 10 και 11, πολύ περισσότερο αυτό είναι, αυτό είναι το χοντρό κομμάτι των εξοπλισμών. 70% ε, και πλέον των εξαγωγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να πουλήσει πολύ σημαντικές ποσότητες όπλων, ας πούμε ε, κανόνια με ε, όλμους, βόμβες, τορπίλες, πύραυλους, κατηγορία 4 ή ε, πολεμικά πλοία, ε, υποβρύχια, κατηγορία 9, αεροσκάφη στρατιωτικά, έχουμε και πολεμικά αεροπλάνα, κατηγορία 10 και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στρατιωτικής φύσεως, η κατηγορία 11. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ε, όπλων, οι προφορίες που έχουμε μας δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά όπλα το 2015 φτάσανε σε δύο βασικούς τομείς. Σας είπα ότι επικεντρωθήκαμε στο 2015. Ε, το 24% είναι ε, τα μεγάλα πλοία και αεροσκάφη. Είχαμε το 24% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το, το, τον προορισμό αυτών των εξοπλισμών, είχαμε Τέσσερις από τις δέκα άδειε εξαγωγών ε, σε απόλυτη τιμή ε, πήγαν στην ε, Μέση Ανατολή. Δηλαδή, εγκρίθηκαν κάποιοι εξοπλισμοί το 2015 για εξαγωγές όπλων, έτσι, από τα κράτη-μέλη και τα περισσότερα από αυτά τα όπλα πήγαν στη Μέση Ανατολή, που είναι μια περιοχή όπου πραγματικά υπάρχουν προβλήματα ως προς τη φύση των συγκρούσεων. Επιπλέον, Έφτασε και το 29% ε, αεροσκαφών και άλλων όπλων από την Ευρώπη. Βλέπουμε την τάση προς την οποία κινείται η αγορά. Ε, επίσης, ε, στην, νοτιοανατολική Ασία ε, περνάει εκεί σημαντικό κομμάτι των εξοπλισμών Έχουμε αύξηση των αδειών για εξαγωγές προς τα εκεί, 15 ε, και 17%. Πολλοί στρατιωτικό εξοπλισμό πηγαίνουν λοιπόν στην Ασία. Με βάση λοιπόν την ε, χρονική εξέλιξη που κάναμε, τη χρονική εξέλιξη και την ανάλυση που κάναμε από το 2010, 2003 μέχρι το 2015, βλέπουμε ότι οι ανταλλαγές όπλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, μειώνεται. Και η Ένωση εξάγει όπλα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι η τάση. Ε, βλέπουμε αυτή την τάση, ας πούμε, ε, και πώς εξελίσσεται, κυρίως προς τη Μέση Ανατολή στέλνουμε όπλα και δευτερευόντως στην Ασία. Με αυτή την πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση για τις τάσεις και τους τόπους όπου εξάγονται τα περισσότερα ευρωπαϊκά όπλα, μπαίνει ένα πρώτο ερώτημα. Με ποιο τρόπο οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν μέσω μιας πολιτικής δυναμικής και με μεγάλη επιτυχία εξαγωγής, ε, στην εξαγωγή όπλων, πώς λοιπόν συνεισφέρει στην ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς συνεισφέρει στην αύξηση της βίας ανά τον κόσμο, γενικά και σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες ειδικά. Και προσπαθούμε να αναλύουμε την επίπτωση που είχε αυτή η μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ευρώπη προς ορισμένες χώρες. Κάναμε μια λεπτομερή ανάλυση, την οποία θα παρουσιάσει ο Μαρία Βιέγιας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρία Βιγέγιας Κυρία Μαρία Βιέγε. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω για τις έρευνε που κάναμε. Ευχαριστώ γι' αυτό, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δούμε το, την πρώτη διαφάνεια που έχουμε ετοιμάσει, αν γίνεται. Το 2015 είναι η χρονιά που, όπως σας είπε ο συνάδελφος, αναλύσαμε. Ε, σε όλο τον κόσμο είχαμε 35 ένοπλες συγκρούσεις διαφορετικής φύσης και με διαφορετικούς βαθμούς στρατιωτικοποίησης και έντασης που προκάλεσαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ασφάλεια και την, τους αμάχους πληθυσμούς. Οι περισσότερες ε, συγκρούσεις έγιναν στην Αφρική και στην ε, Ασία, 13 στην Αφρική, 12 στην Ασία, ενώ στη Μέση Ανατολή είχαμε 6 ένοπλες συγκρούσεις, στην Ευρώπη 3 και στην Αμερική 1. Από τις 35 ένοπλες συγκρούσεις που είναι, διαπιστώσαμε το 2015, ε, αυτές έλαβαν χώρα σε 27 χώρες. Από αυτά τα 27 κράτη, 13 βρίσκονται μεταξύ των 50 πιο σημαντικών χωρών εισαγωγέων όπλων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίγυπτος, Ινδία, Τουρκία, Ιράκ, Ταϊλάνδη, Αλγερία, Πακιστάν, Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ, Ουκρανία, Νιγηρία και Κολομβία με φθήνουσα σειρά, αν με βάση τον όγκο εισαγωγών. Από αυτέ τι 13 χώρε που σα ανέφερα, είχαμε εκεί 16 ένοπλε συγκρούσει. Γιατί σε ορισμένε από αυτέ είχαμε περισσότερε από μία ένοπλε συγκρούσει ε, την ίδια στιγμή, όπω παραδείγματο χάρη στην Ινδία, με τι ε, επιθέσει στο Ασάμ, στο Χάμου και στην Κατσεμίρα ε, και με την σύγκρουση με, την, με τη μαοιστική οργάνωση CPIM, καθώς και στο Πακιστάν ε, που είχαμε σύγκρουση μεταξύ Ταλιμπάν και κράτους, ε, πακιστανικού κράτους και στον Παλουτσιστάν. Ε, στο 2015 σε 31% από αυτές τις συγκρούσεις είχαμε υψηλά επίπεδα βίας. Το επίπεδο θνησιμότητας ξεπέρασε τα, τους χίλιους νεκρούς το χρόνο και μερικές φορές κατά πολύ. Πέντε από τις 11 συγκρούσεις υψηλής έντασης το 2015 έγιναν σε χώρες που βρίσκονται μεταξύ των 50 πιο σημαντικών χωρών εισαγωγέων ευρωπαϊκών όπλων, ε, όπως η Νιγηρία, το Πακιστάν, η Ουκρανία, η Αίγυπτος και το Ιράκ. Μεταξύ αυτών πρέπει να τονίσουμε τον πόλεμο στο Ιράκ που προκάλεσε τουλάχιστον 17.578 ε, νεκρούς το 2015. Σε πολλούς από αυτούς τους ε, πολέμους πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε επίπεδα βίας ε, που αυξήθηκαν μετά το 2015. Από την εποχή δηλαδή που επισημοποίησαμε, τυποποίησαμε ας πούμε, τον τρόπο πώληση όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το, η Τουρκία, το Ιράκ, στην πακιστανική επαρχία του Μπαλουτσιστάν, στο Χάμου και στην Κατσεμίρα και στην ε, σύγκρουση ε, που φέρνει που στη μαγιστική οργάνωση PIM ε, με την Ινδία. Σε ορισμένε περιπτώσει όπω στην Τουρκία και στην Ινδία η κλιμάκωση της βίας ε, έφτασε το μέσο ή το υψηλό επίπεδο. Το 2015 η σύγκρουση στην Ινδία είχε κατηγοριοποιηθεί ως χαμηλής έντασης ενώ της Τουρκίας ως μέτριας ένταση Λόγω πέρα από τα θύματα προκαλούν, οι συγκρούσει αυτέ το 2015 είχαν σοβαρότατε επιπτώσει στον πληθυσμό. Ε, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλήματα στην ανθρώπινη ασφάλεια. Μεταξύ των συνεπειών τη βία ε, πρέπει να τονίσουμε την υποχρεωτική μετακίνηση πληθυσμών. Στα τέλη του 2015. Ποιο... Τόσο μικροφόνο συζήτηση. Σα μπερδέψαμε λιγάκι. Γιατί η κυρία Κλειφ μιλούσε αρκετά αργά προηγουμένω. και παρόλα αυτά ε, λάμβανα μηνύματα ότι μιλάει πολύ γρήγορα και τώρα ακούω κάτι που ε, το προφέρει η κυρία τρομερά γρήγορα. Σας παρακαλώ, λίγο πιο αργά. <clears throat> Στα τέλη του 2015 είχαμε 65,3 εκατομμύρια άτομα τα οποία ε, υποχρεωτικά μετατοπίστηκαν με βάση τον απολογισμό της ΑΚΝΟΥΡ. Αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι εκτοπιστέντες πληθυσμοί διπλασιάστηκαν. Ε, η Κολομβία είναι μία από τις 10 πρώτες χώρες που παράγουν πρόσφυγε σε παγκόσμιο επίπεδο και βρίσκεται στον κατάλογο των 50 πιο σημαντικών χωρών που εισάγουν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα νούμερα των ε, προσφύγων από την Κολομβία έφτασαν στις 340.000 και πλέον στα τέλη του 2015. Επιπλέον, χώρες που εισάγουν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται μεταξύ εκείνων που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό εκτοπιστέντων ανθρώπων ε, το 2015, το, όπως η Κολομβία, το Ιράκ, η Νιγηρία και το Πακιστάν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την προοπτική του φύλου και τις επιπτώσεις που έχουν οι, πόλεμοι στη βία στις γυναίκες. Μπορούμε να τονίσουμε ότι 7 από τις ε, ε, συγκρούσεις που έγιναν σε χώρες που βρίσκονται μεταξύ των 50 πιο σημαντικών χώρων που εισάγουν όπλα από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επίπεδα ε, διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου πολύ ψηλά. Ιράκ, Ινδία, Ινδία, Πακιστάν και Νιγηρία με βάση τον, ε, τα όσα λέει όσα. Επιπλέον, τρεις ένοπλες συγκρούσεις που έγιναν ε, σε χώρες οι οποίες βρίσκονται στις, στον κατάλογο των 50 χωρών ήταν θέατρα σεξουαλικής βίας που συνδέονται με την ένοπλη σύγκρουση. Αναφέρετε τόσα πολλά νούμερα με τόσο γρήγορο τρόπο που δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. The Να περάσει το μήνυμα. Συγγνώμη. <clears throat> Τρεις ένοπλες συγκρούσεις που έγιναν σε χώρες που βρίσκονται σε αυτό το κατάλογο των 50 χωρών που εισάγουν τα περισσότερα πολλά όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν θέατρα σεξουαλική βία που συνδέονται με, την, με τον πόλεμο, με την ενοπλή σύγκρουση, με, βάση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το 2015. Και είναι η Κολομβία, η Νιγηρία και το Ιράκ. Όπω ε, υπόθηκε και προηγουμένω, η κοινή θέση δεν αναφέρει αποκλειστικά την κατάσταση ένοπλης ε, σύραξης αλλά αναφέρεται γενικά ε, και σε χώρες που υπάρχουν εντάσεις. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι το 2015 20 από τις 50 βασικότερες χώρες που εισάγουν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε μια τέτοια σως κοινωνικοπολιτική κατάσταση έντασης όπως το Μαρόκο, η Νιγηρία, Μεξικό, Περού, Νότια Κορέα, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Ουσμπεκιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ρωσία, Σερβία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ιράκ, Ισραήλ και Λίβανος που μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε πρόβλημα εκεί. αυτές οι 20 χώρες αντιμετώπισαν 29 διαφορετικά είδη εντάσεων. Μερικές από αυτές τις εντάσεις είχαν διεθνή χαρακτήρα. Τρεις από τις πέντε βασικές ε, χώρες που εξάγουν όπλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσταν θέατρο εντάσεων ε, το 2015, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Ινδία. Η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός προορισμός ε, ευρωπαϊκών όπλων. Πρόκειται για μια περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική δεδομένη της ε, στρατιωτικής θέση και παρέμβαση της Σαουδική Αραβίας στη σύγκρουση τη Ιεμένης το 2015 που ε, δημιούργησε και εσωτερική αστάθεια στην ίδια την ε, Σαουδική Αραβία. 9 από τις 18 ε, περιπτώσεις ε, έντασης υψηλής ε, κλίμακας το 2015 βρισκόταν σε χώρες που ε, έπαιρναν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιγηρία, Ινδία, Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ρωσία, Αίγυπτος, Ισραήλ και Λίβανος. Δηλαδή, πρόκειται για εντάσεις με σημαντικό επίπεδο βίας και ή πολιτικά και κοινωνικά κινήματα ας και εντάσεις πολύ σημαντικές. Επιπλέον, επιπλέον εννέα χώρες ε, όπου είχαν εντάσεις στο εσωτερικό τους είχαν παράλληλα και πολέμους το 2015. Η Νιγηρία, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Ταϊλάνδη, η Ρωσία, η Αίγυπτος το Ιράκ και το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα σύνολο 12 ενοπλών σειράξεων. Και η κατάσταση ε, αυτών των χωρών ήταν ιδιαίτερη σε ό,τι αφορά την, ε, τη βία. Δηλαδή πέρα από την ε, ένοπλη σύραξη είχαμε και βία και πολιτική βία. Διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν εντάσεις και εισάγουν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν και τεράστιο αριθμό εσωτερικά εκτοπιστέντων το 2015, όπως το Ιράκ, η Νιγηρία και το Πακιστάν. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επίπτωση στο φύλλο, πρέπει να τονίσουμε ότι 7 από τις χώρες που έχουν κοινωνικοπολιτικές εντάσεις, ε, που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες ε, ανήκουν σε αυτόν τον κατάλογο των 50 πιο σημαντικών χωρών που παίρνουν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν σε χώρε όπου έχουμε υψηλή διακριτική μεταχείριση ανάμεσα σε άντρε και γυναίκε. Με βάση με τον δείκτη για την ανισότητα των φύλων του ΟΗΕ. Νιγηρία, Ινδία, Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Αίγυπτο, Ιράκ και Λίβανο. Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι οι ευρωπαϊκέ εξαγωγέ όπλων πήγαιναν σε προορισμούς που ε, και σε χώρες όπου βρίσκονται σε ένοπλη ή σε ένταση. Αυτό παραβιάζει κατάφορα την κοινή θέση σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ε, τεχνολογικού, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτικής τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι το εμπόριο όπλων δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση πολιτική που επιτείνει τις ενόπλες συγκρούσει και σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κριστόφ Κριστόν της Γκριπς. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε σωθόνες την παρουσίασή μου. Θα ξεκινήσω και θα ακολουθήσει η παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα προσεστώ. Κριστοφό Στιερνών το όνομά μου, είμαι ερευνητή στο GRIP, είναι η ομάδα για έρευνα και ενημέρωση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Από εκεί βγαίνει το GRIPS. Είμαστε ομάδα προβληματισμού που εδρεύει στι Βρυξέλλε για θέματα ειρήνη και ασφαλεία. Το έργο μου καλύπτει την μετακίνηση ε, όπλων, έλεγχο εξαγωγή όπλων, μικρά όπλα, ελαφρύ οπλισμό. Κατά τη διάρκεια του επόμενου δεκαλέπτου θα επικεντρωθώ επί προσφάτων περιφερειακών τάσεων ε, για τα θέματα των μεταφορών όπλων. Οι περισσότερες πληροφορίες που θα σας παρουσιάσω προέρχονται από το έργο του ΣΥΠΡΙ. Είναι το Διεθνές Ινστιτούτο για την Έρευνα την Ειρήνη που εδρεύει στη Στοκχόλμη τα στοιχεία από τη Σύπρη αφορούν τη μεταφορά μεγάλου όπλων, μαχητικών αρισκοφών ελικοπτέρων, θωρακισμένων οχημάτων, συστήματα μεγάλου διαμετρήματος. Εξαιρούνται τα μικρά και ελαφρά όπλα και τα πυρομαχικά αυτών, όλα τα υπόλοιπα. Τώρα για το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έρευνα, ιδιαίτερα σήμερα που ο όγκος των διεθνών μεταφορών μεγάλων όπλων αυξάνεται σταθερά για περίπου 15 χρόνια. Όσο όγκος παραδόσων μπορεί να διακυμαίνεται κάθε χρόνο, η σύπρη μας παρουσιάζει στοιχεία για μια πενταετή περίοδο, για πενταετής περίοδους και έτσι έχουμε μια πιο σταθερή αποτύπωση των τάσεων. Από το 2013 με το 2017 ο όγκος των διεθνών μεταφορών των μεγάλων αυτών όπλων ήταν 10% υψηλότερος από την προηγούμενη πενταετία. Κατά την τελευταία πενταετία το Τσίπρι ε, ενετόπισε 67 χώρες ε, ως εξαγωγής ε, μεγάλων όπλων. Η αγορά εξαγωγής όπλων είναι πολύ συγκεντρωμένη αγορά με περίπου 75% των συνολικών όγκων εξαγωγών όπλων στα χέρια πέντε χωρών και μόνο. Οι μεγαλύτεροι είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, ακολουθεί η Ρωσία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Κίνα. Και αυτές οι πέντε χώρες έχουν αυξήσει το συνολικό μερίδιο της αγοράς με την πάρα του χρόνου με συνδυασμένες εξαγωγές που αυξάνουν ταχύτερα από το σύνολο. Οι, πάνω οι, οι πιο σημαντικές χώρες εξαγωγών καλύπτουν το 90% των εξαγωγών όπλων. Τα στοιχεία του ΣΥΠΡΙ ε, δείχνουν σαφώς ότι οι χώρες εκτός ε, της Ευρώπης και Βορείου Αμερικής διαδραματίζουν μικρό ρόλο στις εξαγωγές όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τις πιο σημαντικές 10 χώρες, οι 6 είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις 25 πιο σημαντικές χώρες οι 10 είναι ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Οι πέντε μεγαλύτεροι εξαγωγείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία. Από το 2008 μέχρι το 2012 και το 2013 μέχρι το 2017 οι εξαγωγές όπλων από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27% και του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 37%. Οι εξαγωγές όπλων τη Γερμανία αντιθέτως μειώθηκαν κατά 14%. Οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν ο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων και κατά πολύ με 34% του συνόλου και η Ρωσία παραμένει στη δεύτερη θέση με 22%. Αλλά συνδυασμένε εξαγωγέ από τα κράτη με τη Ευρωπαϊκή Ένωση των όπλων ήταν 27% του συνολικού ε, συνολικών εξαγωγών στον κόσμο την τελευταία πενταετία και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη όπλων ε, πριν τη Ρωσία, πάνω τη Ρωσία. Ε, η Μέση Ανατολή είναι ο βασικός προορισμός των ευρωπαϊκών όπλων. Οι γερμανικές εξαγωγές κυρίως πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ασία και Οκεανία είναι η επόμενη βασική προορισμοί των ευρωπαϊκών όπλων. Ας ρίξουμε μια ματιά και να δούμε που πηγαίνουν τα αμερικανικά όπλα. Οι αμερικανικές εξαγωγές είναι οι μεγαλύτερες. Εξα... Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 25% στην περίοδο 2008-2012 και 2013-2017. Έτσι δε περαιτέρω αυξήθηκε το χάσμα με τις άλλες σημαντικές εξαγωγικές χώρες. Εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ το 2017 ε, ήταν οι μεγαλύτερες μετά το 1998 οι ΙΠΑ παρέδωσαν μεγάλα τέτοια όπλα σε τουλάχιστον 19 διαφορετικές χώρες κατά τελευταία πενταετία και από τους 50 μεγαλύτερους αγωγείς στον κόσμο όπλων μόνο οι 7 ε, εισαγωγείς δεν έλαβαν όπλα από τη ΣΥΠΑ. Η Σαουδική Αραβία είναι κατά πολύ ο μεγαλύτερος αποδέκτης των Αμερικανικών όπλων με αύξηση 448% κατά την περίοδο που αναφέρουμε. Οι ΙΠΑ επίσης αύξησαν, βελτίωσαν τις ε, σχέσεις με την Ινδία με αύξηση πάνω από 500% με την πάροδο των ετών. Η Ρωσία ε, οι εξαγωγές της Ρωσίας μειώθηκαν κατά 7,1% κατά την καλυπτόμενη περίοδο και η Ρωσία εξήγαγε σε 47 χώρες με την Ινδία, την Κίνα και το Βιετνάμ μαζί να δέχονται το 58% όλων των ρωσικών εξαγωγών όπλων. Τώρα πέρα από τις πέντε πιο σημαντικές χώρες που εξάγουν όπλα τα στοιχεία του ΣΥΠΡΙ έδειξαν σημαντικές εξελίξεις σε άλλε χώρε που εξάγουν όπλα, μεγάλες αυξήσει εξαγωγέ όπλων από το Ισραήλ, την Νότια Κορέα και την Τουρκία. Η Νότια Κορέα εξήγαγε στις ευρωπαϊκές χώρες για πρώτη φορά όπλα κατά την καλυπτόμενη περίοδο και η Τουρκία αυξήσει σημαντικά εξαγωγέ όπλων προ άλλε χώρε τη Μέση Ανατολή. Πού προέρχονται είδαμε τα όπλα, πού έρχονται τα όπλα, ας δούμε τώρα πού πήγανε τα όπλα και πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Κατά την περίοδο 2013-2017, 42% των εισαγωγών αυτών των μεγάλων όπλων ήταν στην Ασία και την Οκεανία. Αυτό, αυτός ήταν ο προορισμός. Ακολουθεί η Μέση Ανατολή με 32%, η Ευρώπη, η Αφρική ε, και η Αμερικανική Ήπειρος. Λοιπόν, οι εισαγωγέ όπλων από χώρε Μέση Ανατολή αυξήθηκαν πάνω από 100% κατά την καλυπτόμενη περίοδο και κατά 1,8% στην Ασία και Οκεανία. Αντιθέτω, όλε οι άλλε περιοχέ ε, σημείωσαν ε, μείωση των εισαγωγών, μείωση μεγαλύτερη του 20%. Δεν μας εκπλήσει το ότι οι πέντε μεγαλύτερες εισαγωγείς αυτών των μεγάλων όπλων βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και την Ασία, ξεκινώντας από την Ινδία, Σαουδική Αραβία μετά, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κίνα. Μαζί αυτές οι πέντε χώρες αποτελούσαν 35% των συνολικών εισαγωγών αυτών των μεγάλου όγκου ε, όπλων. Μέση Ανατολή, περίπου το 5% του πληθυσμού του κόσμου έχει η Μέση Ανατολή, αλλά απορρόφησε περίπου το 1 τρίτο όλων των εισαγωγών όπλων στην περίοδο 2013 μέχρι 2017. Τα πρόσφατα έτη οι περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής ενεπλάκησαν άμεσα σε βίες συγκρούσεις. η στρατιωτική παρέμβαση στην Ιεμένη είναι η πιο σημαντική απόδειξη μέχρι τώρα της μεγαλύτερης προθυμίας και δυνατότητας των αραβικών κρατών να χρησιμοποιούν τις μεγάλες ποσότητες εισαγωμένων όπλων εκτός των δικών τους ε, συνόρων. Η Σαουδική Αραβία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων σε όλο τον κόσμο, είναι και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας της περιοχής με 31% των συνολικών εξαγωγών της περιοχής. Ακολουθεί η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ιράν, παρόλο που το πιο έχει τον περισσότερο πληθυσμό στη Μέση Ανατολή, είχε μόνο το 1% των εισαγωγών στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα μισά όπλα που μετεφέθησαν στη Μέση Ανατολή προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Από τις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή όπλων, όλες εκτός από μία έχουν κάποια εξάρτηση από τις εξαγωγέ όπλων προς τη Μέση Ανατολή. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Φιλανδία όλες έχουν μία ή περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής ε, ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους πελάτες τους. Άλλες χώρες όπως είναι το Βέλγιο που είναι εκτός της μελέτης διότι εξάγει κυρίως μικρά όπλα και ελαφρά όπλα ε, δείχνουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και εδώ θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. που ήρθατε στην συζήτησή μας. Πριν ε, δώσω τον λόγο στους ε, συντονιστές, ε, δράτω με τις ευκαιρίες και εγώ να κάνω κάποια σχόλια και να ρωτήσω τους κυρίους Στερνών και Βιλέγιας. Αναφέρατε, κυρία μου, την Ουκρανία και πόσο κατάλαβα ε, και μπορεί βεβαίως να μην μεταφέρθηκε ακριβώς γιατί μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα ακούγα εγώ τα αγγλικά Αναφέρατε λοιπόν την Ουκρανία. Η ε, κυρία μου, η Ουκρανία πράγματι έχει μια σύγκρουση. Δεν υπάρχει εμφύλιος όμως. Δεν είναι ενδοκρατική η σύγκρουση. Ε, πρόκειται για επίθεση από το εξωτερικό και παράνομη προσάρτηση. Και για τα δεδομένα του κυρίου Στερνών ότι στην ε, περίοδο αυτή είχαμε μείωση των ρωσικών εξαγωγών πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, το ότι είχαμε τεράστια ροή ρωσικών όπλων στην Ανατολική Ουκρανία και βεβαίως ε, στην ε, προσαρτημένη Κρυμαία. Ξέρω ότι είναι στατιστικά στοιχεία αυτά, αλλά όταν μιλάμε βεβαίως για τόπους ε, συγκρούσεων, ε, είμαστε πολιτικοί που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Επίσης είμαι κάπως περίεργη για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν ε, το Ιράν, ε, γιατί υπήρχαν φήμες για το ότι δεν ε, είχαν καταγραφεί σωστά οι παραδόσεις ρωσικών όπλων στο Ιράν. Η ερώτησή μου λοιπόν, ε, η γενική αφορά τις παραδόσεις όπλων που δεν καταγράφονται και η πιθανή ανιχνευσή τους ε, με βάση την ε, φύση της σύγκρουσης. Και στη Συρία προφανώς Λοιπόν, να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Τον λόγο έχει ο κύριος Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση απευθύνεται στην κυρία Κλειφ ως ε, συμπρόεδρο. Ε, εσείς ε, προεδρεύετε βεβαίως στην Επιτροπή όπου θα αξιολογηθεί η κοινή θέση. έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση γιατί γνωρίζω ότι στην σύμβαση των κυβερνητικών εταίρων στη Γερμανία είπαν ότι θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω το θέμα. Έχετε λοιπόν δει κάτι από πλευράς ε, Γερμανίας προς ποια κατεύθυνση δηλαδή θα αναπτύξουν το ζήτημα την ε, κοινή θέση και ειλικρινά δεν έπιασα την ε, σύνδεση μιλήσατε για τη μεταχείριση των γυναικών και την σχέση με τις εξαγωγές όπλων η ιδιαιτερότητα δηλαδή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των γυναικών και η σχέση με τα όπλα. Εισαγωγή, εξαγωγή δεν είχα καταλάβει. Ε, επί της ουσίας βεβαίως οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση ε, εις βάρος των γυναικόπαιδων εντάξει αλλά δεν κατάλαβα τη σχέση λοιπόν Τώρα δεν ξέρω βεβαίω, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έφταιγε και η διαμηνία. Λοιπόν, είναι ενδιαφέροντα επίση τα στατιστικά σα στοιχεία, κύριε Στιαρνό, για το ποιοι είναι οι εξαγωγεί ε, και οι εισαγωγεί. Και οπωσδήποτε θα θέλαμε να δούμε σε ποιου τομεί ή θα έπρεπε να είναι σαφές Πού πάνε οι εξαγωγές. Γιατί έχει διαφορά όταν μια χώρα του ΝΑΤΟ στέλνει όπλα σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό εξαγωγή είναι. Ή εάν ε, τα ίδια πήγαιναν ε, σε μια σύγκρουση. Δηλαδή αν μια χώρα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη να γίνει η διάκριση μεταξύ εξαγωγών σε άλλες χώρες ε, της Ένωσης ε, και του ΝΑΤΟ ή ας πούμε έτσι παρόμοιες Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία. Εάν μπορούμε να το υπολογίσουμε χωριστά κάτι τέτοιο, νομίζω ότι έτσι θα είχαμε περισσότερα στοιχεία πιθανής ε, αποσταθεροποίησης ή σύγκρουσης γιατί δεν νομίζω ότι εάν η Πολωνία κάνει εξαγωγή στη Γερμανία ή το αντίστροφο υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια σύγκρουση αλλά αν μια χώρα στείλει απευθείας ε, κάτι σε μια εμπόλεμη χώρα ε, εντάξει μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο οπότε υπάρχει ίσως κάποιος τρόπος να γίνει πιο διαφανής η κατάσταση για να πούμε ότι ε, ενισχύουμε κάποιες συγκρούσεις ή όχι και να διακρίνουμε από τις εξαγωγές σε συμμάχους. Ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις. Ε, ναι, να περιμένω. Για αυτό το οποία μας είπατε. Εγώ είμαι εισηγήτρια φέτος ε, για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της ε, ΣΕΝΤΕ για τις ευρωπαϊκές ε, εξαγωγές όπλων και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Κάλβο και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια πολιτική διάσταση Δηλαδή, το τομέας ε, της εξαγωγής όπλων είναι ένα θέμα αντιφατικό. Δηλαδή υπάρχει η αντίφαση μεταξύ της ε, κοινωνικής αποδοχής ε, και της πραγματικότητας. Δηλαδή, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει συνένεση ε, κατά των εξαγωγών όπλων και ειδικά σε περιοχές ε, κρίσης και μετά βλέπουμε πως έχει η πραγματικότητα. Και υπάρχουν οι διάφορες ε, απαιτήσει και οι διαφορές δηλαδή μεταξύ της κοινή θέσης της Ένωσης και της πραγματικότητας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη Σαουδική Αραβία μια χώρα στην οποία η, η οποία συνεχώς είναι στα ΜΜΕ και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση και βεβαίως γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται τα όπλα σε συγκρούσεις και ταυτόχρονα έχουμε αυτόν τον ε, ισχυρό ρόλο των εξαγωγών ε, προς την ε, Σαουδική Αραβία. Οπότε τι πρέπει να βελτιώσουμε στο πολιτικό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή με την ε, πραγματικότητα και το ερώτημά μου προς ειδικούς είναι ποια συμπεράσματα θα βγάζατε εσείς, ε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί για να υπάρξει ακριβώς ε, μια μεγαλύτερη ικανοποίηση του κοινού αισθήματος. Μετά ακούσαμε ότι έχουμε το EDPD, το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βιομηχανικό Πρόγραμμα, κάτι το οποίο βεβαίως μπορεί να είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και εκεί πέρα το ερώτημά μου είναι εάν ε, οι ειδικοί τα έχουν ε, συμπεριλάβει αυτά στα συμπεράσματά τους. Το πώς ε, δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις και αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Και κύριε Γκαλέρε, ε, μπαίνω στον πειρασμό να απαντήσω και εγώ μόνη μου στην ερώτησή σας. Δηλαδή το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών σε κάποιες χώρες είναι δείκτης, θα έλεγα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώ. Ας ε, θυμηθούμε πώς ήταν η κατάσταση στο Αφγανιστάν ε, που ήταν ακριβώς ε, κάτι το οποίο ήταν και κίνητρο και εξήγηση της παρέμβασης στο Αφγανιστάν. Και εκεί πέρα νομίζω έχουμε μια σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης της κατάστασης μιας χώρας και της κατάστασης των γυναικών. Βεβαίω, εντάξει, τώρα πλέον κανείς δεν ενδιαφέρεται για το αν η παρέμβαση βελτίωσε την κατάσταση των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βαλέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλα αυτά είναι καταθλιπτικά όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνεται, παρότι τις ξέρουμε, μας καταθλίβουν. Όταν βλέπουμε τα νούμερα τόσο σαφώς, πραγματικά υπάρχει μία θύπνιση. Υπάρχει πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε στην τηλεόραση και στα δίκτυα ότι τα ευρωπαϊκά όπλα πέφτουν σε λάθος χέρια, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Αλλά και αλλού. Υπάρχει πρόβλημα που μας με το σύστημά μας κάπου αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κοίταξα την εκθεσή σας. Τις εκθέσεις από το Πανεπιστήμιο ΠΑΟΥ της Βαρκελόνης. Και την κατάσταση σε διάφορες χώρες για το 2015. Η Γαλλία έχει 36% όλων των εξαγωγών. Παράλληλα, έδωσαν άδειε. 77% όλων των εξαγωγών όπλων το 2015 πήρε άδειε. Παράλληλα, ξέρουμε ότι πάρα πολλά πράγματα που εξάγονται και παίρνουν άδεια για να εξαχθούν πάνε στη Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία κτλ παρότι υπάρχουν πόλεμοι, παρότι υπάρχουν σειράξει ή σειράξει στι οποίε εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία, όχι εντό Σαουδική Αραβία, δηλαδή εκτό. Ε, με βάση τα κριτήρια δεν θα έπρεπε να δώσουμε αυτέ τι άδειε για εξαγωγέ όπλων, γιατί είναι χώρε, ε, πάνε σε χώρε που βρίσκονται σε ενόπλη σύραξη. Είναι εναντίον τη κοινή θέση. Πώ ε, συνδυάζονται, πώ ε, μπορούμε να δεχτούμε αυτέ τι εξαγωγέ και παράλληλα να έχουμε και την κοινή θέση που μιλάει για κάποια κριτήρια. Ε, το 77% του μεριδίου της Γαλλίας αφορά όλες τις εξαγωγές. Όταν δούμε όλα τα ποσοστά, ας πούμε, για τη Συνταγωγική Αραβία ή για τη Μέση Ανατολή, βέβαια δεν διάβασα όλη την έκθεση ακόμα, που έχει και πάρα πολλά στοιχεία, λέει κάπου η έκθεση για τη χώρα μου, με τη Σουηδία, ότι υπήρχε μια μείωση στις εξαγωγές της Σουηδίας. Νομίζω ότι αυτό μας λέει ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί, αν όχι γενικά η κοινή γνώμη στη Σουηδία, η οποία είναι κατά των εξαγωγών όπλων. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε νομοθετικές αλλαγές. Ε, στις 14 Απριλίου μάλιστα αλλάξαμε τον νόμο για την πώληση όπλων και ο νόμος αυτός προβλέπει πολύ πιο αυστηρά κριτήρια για να εξάγουμε σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Ε, κοινή γνώμη τροφοδοτεί και μία νομοθετική αλλαγή και αντίστροφα. Επίσης Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, ε, Εμμυράτα ε, είχαν τελείως διαφορετικά μερίδια πριν από περάσει αυτός ο νέος νόμος. Ίσως αλλάξουν οι στατιστικές μας λοιπόν μετά τον νόμο αυτό. Βλέπετε άλλες χώρες όπου το θέμα της κοινή γνώμης μπορείς να, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί δηλαδή να οδηγήσει σε αυστηρότερη νομοθεσία για την ε, εξαγωγή όπλων. Η νομοθεσία η οποία να προβλέπει ότι οι χώρες οι οποίες εξάγουμε όπλα θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της κοινή θέση. Ελπίζω να, με καταλάβατε. Δεν ξέρω από την ε, έκφρασή σας αν τα καταλάβατε όλα, αλλά ελπίζω καταλάβατε. Αλλιώ θα σα το πω ισπανικά. Ο κύριο Λίτ, σα ε, σας ευχαριστώ για τι παρουσιάσει σα. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε ο κύριο Γκάλερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε ε, για τους προορισμούς των εξαγωγών όπλων. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο για τη διπλή χρήση. Ε, το ξέρετε, το έχετε λάβει υπόψη σας στη δουλειά σας. Το έχουν συμφωνήσει αυτό το πλαίσιο οι βουλευτές. Τώρα έχει πάει στη δεύτερη φάση. Τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα. Επίσης, να σταματήσουμε τα εργαλεία βασανισμού. Δεν θα πρέπει να εξάγονται. Ε, απαγορεύονται να εισάγονται. Έχετε στοιχεία για εταιρείε όπου έχουν γραφεί, ας πούμε, αλλού στον κόσμο, ούτως ώστε να μπορούν να παρακάμπτουν τις, τα δικά μας τα εμπόδια. Ξέρετε το πρόβλημα αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και πώς θα επηρεάσει εξαγωγές όπλων. Δεύτερον, τι άποψη έχετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί συζητάμε τώρα το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Το Κοινοβούλιο λοιπόν πώς μπορεί να παίξει ένα ρόλο και στο θέμα των εξαγωγών όπλων. Φυσικά αυτό το θέμα έχει να κάνει με, την, με τα κράτη-μέλη. Ε, θα παραμείνει η αρμοδιότητά του στο θέμα των όπλων. Αλλά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποιος θα μπορούσε να είναι ή ποιος πρέπει να είναι. Ευχαριστώ. Ήταν η ποιο πρεπει να ειναι ευχαριστω παρέμβαση και τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές του πάνελ για να απαντήσουν. Ο καθένας από εσάς έχει 6 λεπτά ή 5 λεπτά question post or eventual additional remarks. We start with Mrs. Cliff. Ξεκινάμε την κυρία Κλίφ. Ε, thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους έθεσαν ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα που απευθύνθηκε ήταν από τον κύριο Γκάλερ. Πράγματι, από τα κράτη-μέλη η Γερμανία είναι πολύ δραστηριοποιημένη ε, στον αφορά την ομάδα εργασίας. Έχουμε τακτικές ανταλλαγές απόψεων ε, γύρω στους για τους προορισμούς ε, που πηγαίνουν τα όπλα σε κάποιες χώρες. Η Γερμανία πάντα παρέχει πληροφορίες για τα άλλα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ενεργή η συμμετοχή της Γερμανίας Όσον αφορά την κοινή θέση, οι συζητήσεις στην ομάδα εργασίας μόλις ξεκίνησαν. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα. Όμως υπάρχει άτυπη συνεννόηση στην ομάδα, δηλαδή ίσως δημιουργήσουμε κάποιες ομάδες κρούσης συγκεκριμένα θέματα που θα μπορούσαν να προωθηθούν από κάποιο κράτος μέλος. Η Γερμανία έχει εκφράσει ενδιαφέρον Πιστεύω ότι γνωρίζει το παρόν κλίμα και τις συζητήσεις που γίνονται στη Γερμανία και θέλει να συμμετάσχει ενεργά στην ομάδα εργασίας η Γερμανία. Κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις αφορούσαν περισσότερο τους άλλους συναδέλφους στο πάνελ, αλλά με τα χαράς να ξαναλάβω το λόγο αν υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος Ζορδί Κάλβο. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια για τις παρεμβάσεις που άκουσα, για τις οποίες σας ευχαριστώ. Καταρχάς, τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς είναι ανεπαρκή. Πρέπει να τα βελτιώσουμε προφανώς, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν δίνουν πληροφορίες ή δίνουν διαφορετικές πληροφορίες στην εθνική έκθεση από την ευρωπαϊκή. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τα στοιχεία φτάνουμε σε συμπεράσματα που είναι απογοητευτικά, που προξενούν κατάθλιψη, όντως. Υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο για την εξαγωγή των όπλων. Και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει όλο και περισσότερο σε όλο και περισσότερε χώρε, δημιουργώντα μεγαλύτερη ανασφάλεια και περισσότερε συγκρούσει. Αυτό είναι πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που παράγει πραγματικά απογοή... παράγει φαινόμενα ας πούμε, απογοήτευση στον πληθυσμό και χάνει την αξιοπιστία τη. Είναι ευθύνη αυτών που δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ευρωβουλευτών, των πολιτικών, που πρέπει να κάνουν κάτι για να κτίσουν αυτή τη χαμένη αξιοπιστία. Νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, όπως αυτό που έθεσε ο κύριος Γκάλερ, ο οποίος έφυγε όμως, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εκθέσεις ίσως, τα οποία, οι οποίες εκθέσεις θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιοι πουλάνε αυτά τα όπλα σε χώρες ε, όπου η κατάστασή τους επιδεινώνεται ή όπλα τα οποία έχουν πραγματικά αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια. Πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα με ένα ευρωπαϊκό όραμα. Και, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πιο πραγματικό, τίμιο και ανεξάρτητο έλεγχο. Όταν μιλήσαμε με την Ισπανική κυβέρνηση, για αυτό το θέμα, η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση έχει δικές της εσωτερικές ε, εκθέσεις και αξιολογήσεις για να αξιολογήσει αν τα όπλα τα οποία πουλάει ε, καταλήγουν σε λάθος χέρια. Προφανώς θα πρέπει να έχει πολύ καλές εκθέσεις ε, η Ισπανική κυβέρνηση για τη Σαουδική Αραβία και για άλλες κυβερνήσεις που πουλάει όπλα. Πολύ ωραία. Έχετε αυτέ τις πληροφορίε. Α, δώστε μα και εμά λοιπόν. Για να φτάσουμε σε άλλα συμπεράσματα ίσως. Αλλά Χωρίς αυτέ τις ε, ωραίε τις ισορροπημένε εκθέσει, φτάνουμε σε αυτά τα συμπεράσματα που σα ε, παρουσιάσαμε. Επίση, σε 30 δευτερόλεπτα να σα πω ότι είχαμε και μια προηγούμενη έκθεση με αυτή τη λογική. Ε, προσπαθούσαμε να δούμε αν οι εξαγωγέ ευρωπαϊκού εξοπλισμού είχαν επιπτώσει στην ασφάλεια. Λόγω, ας πούμε, παραγωγής ε, προσφύγων ή εσωτερικά εκτοπιστέντων, οι οποίοι τελικά έρχονται και στην Ευρώπη. Και σε αυτή την έκθεση λοιπόν είχαμε δει ότι τουλάχιστον σε 26 προορισμούς μέσα σε 12 χρόνια που πολλούνταν ευρωπαϊκό όπουλα η κατάσταση επιδεινώθηκε ή τουλάχιστον σε καμία περίπτωση η πώληση όπλων δεν βελτίωσε την κατάσταση ε, και σε καμία περίπτωση δεν μειώνονταν ο αριθμός που έφευγε από τις αιστείες του. Αντίθετα, αυξανόταν. Με τέτοιο τρόπο, με τέτοιους δείκτες, φτάνουμε σε συμπεράσματα ότι οι εξαγωγές όπλων από την Ευρώπη έχουν πραγματικά αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια σε πολλές χώρες του κόσμου. Και πιστεύουμε ότι τελικά αυτό συνδέεται και με την ασφάλεια στη δική μας χώρα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εμείς θα πρέπει να ε, ρυθμίσουμε θέματα ανασφάλειας ε, λόγω του ότι συμβαίνει σε ξένες, σε τρίτες χώρες που μας επηρεάζουν. Τώρα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται στον έλεγχο όπλων. Και ποιο είναι αυτό, ότι ο έλεγχος είναι δυνατός γιατί τώρα υπογράφονται συμβάσεις με βάση ε, πιστοποιητικά για τελική χρήση οι χώρες οι οποίες αγοράζουν τα όπλα. Υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, έτσι. Θέλω να καθέσω το εξή ερώτημα. Πώ μπορούμε μετά να δούμε τι συνέχεια δίδεται στη σύμβαση. Πολύ ωραία, υπογράφεται α πούμε. Μετά τι γίνεται. Να ε, κάνει αυτόν τον έλεγχο κάποιο εξωτερικό, ας πούμε φορέας για να δούμε πώ λειτουργεί αυτή η σύμβαση. Έτσι. Γιατί φοβάμαι ότι αυτές οι συμβάσεις ε, υπογράφονται για τα μάτια του κόσμου. Για το Θεαθήνε. Τα όπλα θα πουληθούν. Επίσης υπάρχουν πρωτοβουλίε που βελτιώνουν τον έλεγχο, όπως είναι η περίπτωση τη Σουηδία. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση σε αυτή την περίπτωση. Ίσως η απάντηση λοιπόν είναι ότι τον έλεγχο δεν το κάνει ο ενδιαφερόμενος, έτσι, αν τις ε, εκθέσεις για τον έλεγχο ε, και τις εξαγωγές των όπλων τις κάνει η κυβέρνηση που ξέρουμε πολύ καλά που θέλει να κάνει διάλογο και να κάνει business με, την, με τον κλάδο που πουλάει αυτά τα όπλα, προφανώς αυτές οι εκθέσεις δεν είναι τίμιες και ανεξάρτητες. Εάν θέλει το Κοινοβούλιο να παίξει αυτό το ρόλο, του πραγματικού δηλαδή ελεγκτή μπορεί να έρθει σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, ούτω ώστε να έχει πραγματικά καλά στοιχεία στα χέρια του για να παίρνονται σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρία, η κυρία Μαρία Βιγέγιας. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην ερώτηση για την ε, σημασία της διάστασης του φύλου και των δικαιωμάτων των γυναικών ερώτηση του κυρίου Γκάλερ, ο οποίος έφυγε βέβαια στο μεταξύ. Το, η αρχή της ισότητας των φύλων θα πρέπει να αφορά όλες τις δημόσιες πολιτικές και φυσικά και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας και άρα τελικά και τις εξαγωγές όπλων. Ξέρουμε και διαπιστώθηκε και από τον ΟΗΕ ότι όταν εγκρίναμε την συνθήκη για το εμπόριο όπλων υπήρχε μια συγκεκριμένη ρήτρα για τις επιπτώσεις που έχει το εμπόριο των όπλων στα δικαιώματα των γυναικών. Δηλαδή, η συνθήκη για το εμπόριο των όπλων μας προτρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στις χώρες αυτές όπου εξάγονται τα όπλα. Επίσης, η έκθεση των ΗΠΑ για την αξιολόγηση της κατάστασης των γυναικών και της ασφάλειας το 2015 είπε ότι η στρατιωτικοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο είχε σοβαρότατη επίπτωση στα δικαιώματα των γυναικών. Από διάφορους φορείς και κυρίως από τον ΟΗΕ γίνεται μια προσπάθεια να ληφθεί υπόψη διάσταση του φύλου. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φύλο, η ειρήνη και η ασφάλεια είναι πράγματα συνδέονται, που συνδέονται και προσπαθούμε να συνδέσουμε τα δικαιώματα των γυναικών με την ειρήνη και την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την, τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες αυτές που περνάνε ένοπλη σύραξη, γιατί επιδεινώνουν, επιδεινώνουν τις διακρίσεις εις των γυναικών, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και Επομένως, θα πρέπει να μπουν στο κέντρο τη συζήτηση αυτά τα θέματα όταν μιλάμε για εξαγωγέ όπλων. Τι Thank you, Mr. ευχαριστώ, κύριο κύριος ε, Στιέρνον. Πρώτα απ' όλα θα καλύψω το ζήτημα της ε, διαφοροποίησης ε, των εξαγωγών στα μέλη του ΝΑΤΟ ή τους συμμάχους ε, και τις μη φιλικές χώρες. Δεν έχω ακριβώς ε, τον αριθμό. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από τους 8 μεγάλους εξαγωγείς όλοι τους ε, στους τρεις κορυφαίους πελάτες έχουν τουλάχιστον δύο που δεν είναι μέλη της Ένωσης ή του ΝΑΤΟ ή συμμαχικές χώρες. Οπότε η πλειοψηφία των εξαγωγών πηγαίνουν εκτός ε, χωρών θα τις λέγαμε φιλικές για την διπλή χρήση. Α, δεν εργάζομαι εγώ πάνω στο θέμα, ένα συνάδελφός μου το καλύπτει. Ναι, θα το απαντήσω λοιπόν για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πράγματι θα μπορούσε να αυξηθεί με διάφορους ε, τρόπους. Ε, πρώτα απ' όλα ε, η συζήτηση αυτή αφορά τα διάφορα ταμεία άμυνας. Εάν αρχίσει λοιπόν η χρηματοδότηση αμυντικού εξοπλισμού, το ερώτημα είναι ποια θα είναι η εποπτεία της Ένωσης για την εξαγωγή αυτού του εξοπλισμού. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, στην διαδικασία αναθεώρησης ε, που ανέφερε η κυρία Κλήφε για την ε, κοινή θέση εξαγών ενθαρρύναμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο και ζητάμε από τα νυν ε, κράτη-μέλη να κάνουν αυτή τη διαδικασία με τρόπο ανοιχτό και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα δώσω τον λόγο και πάλι στην κυρία Κλίφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας δώσω κάποια νούμερα όσον αφορά την άρνηση εξαγωγών. Γιατί ε, προφανώς και είναι κατανοητό η Μέση Ανατολή και η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα κλειδί Συγκρίνοντας λοιπόν ε, την 17η, ε, 18η και 19η της έκθεση βλέπουμε ότι είχαμε 6 αρνήσεις αντιστοίχως 7 και μετά ανέβηκαν σε 18 αρνήσεις εξαγωγών στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να μην φαίνονται πολλές αλλά αυξήθηκαν και νομίζω ότι οφείλεται κυρίως ε, στους ευρωβουλευτές και την κοινωνία των πολιτών Όσον αφορά την ε, Μέση Ανατολή συγκρίνοντας την 17η και 18η έκθεση υπήρχαν 14 αρνήσεις εξαγωγών, μετά ανέβηκαν στις 65. Αυτά είναι απλώς κάποια νούμερα. Οι έκθεση είναι στην διάθεσή σας βεβαίως. Κάτι το ενδιαφέρον επίσης ακούστηκε για την σημασία των πιστοποιητικών τελικής χρήσης και να διασφαλίζουμε το ότι τα αγαθά δεν θα πηγαίνουν παραπέρα. Πρώτα απ' όλα βεβαίως είναι μεγάλο ζήτημα όπως είπαμε η παρέκκληση από την πορεία στον τελικό παραλήπτη η διαδικασία πιστοποίησης τελικού χρήστη είναι κάτι το οποίο θα δούμε όταν δούμε την εφαρμογή της κοινής θέσης. αλλά Νομίζω ότι κάποια σχόλια που άκουσα από κράτη-μέλη είναι ότι είναι πρόκληση, είναι θέμα πόρων. Δηλαδή για κάποια κράτη-μέλη ε, δεν έχουν την δυνατότητα όπως οι ΙΠΑ που έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα με το οποίο ελέγχουν που καταλήγουν οι εξαγωγές τους. Για κάποια κράτη-μέλη ίσως υπάρχει θέμα δυνατοτήτων, αλλά κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν. Και ε, θα ήθελα να αναφέρω ένα έργο που στηρίζει η Ένωση, το έργο iTrace, το οποίο είχε αναλάβει ένα ε, οργανισμός που λέγεται έρευνα όπλων και συγκρούσεων. Πηγαίνουν δηλαδή στις περιοχές συγκρούσεων και κοιτάνε τα όπλα και κοιτούν ε, τους αριθμούς τους και από πού προέρχονται και δεν, ε, λένε ελεύθερα από πού προέρχονται, από ποια κράτη-μέλη και ο στόχος είναι να βοηθήσουν ε, τα κράτη-μέλη να έχουν συνέστηση όταν κάνουν αξιολόγηση κινδύνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κάρβερ, έχετε τον λόγο. Κάλβο. Ναι, ε, σύντομα παρακαλώ γιατί έχουμε ολοκληρώσει δυστυχώς. Ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο για να απαντήσω για το θέμα της αλλαγής που υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει περισσότερες ευθύνες για τα θέματα της άμυνας, μια και αφιερώνει όλο και μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού της σε αυτήν. Αυτό συνδέεται με την παρέμβαση της κυρίας Κλίφ για την ε, ικανότητα που έχει η Ένωση να ελέγχει τα όπλα. Είναι το κατά πόσο γίνεται σεβαστή η νομοθεσία η κοινή θέση και όλες, όλοι οι νόμοι που έχουν εγκριθεί στις διάφορες χώρες που εξάγουν όπλα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της πολιτικής βούλησης. Αν η, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανάμε 20 δισεκατομμύρια ας πούμε ε, ευρώ για να προωθήσουμε νέα όπλα, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση, θα πρέπει να υπάρχει μια κριτική, θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, ούτως ώστε να κάνουμε και εκθέσεις και να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των όπλων και να κάνουμε μια συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε όλο αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση σε αυτό το στάδιο. Να σας υπενθυμίσω ότι παρά τις ηλυμένες αποφάσεις οι περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και είναι τομέας του Συμβουλίου βασικά. Βέβαια, αλλάζουν, προδεύουν τα πράγματα και παρακολουθούμε τα εκτενόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους ομιλητές μας. Ευχαριστούμε, διακόπτουμε και καλή σας όρεξη. Like to remind you that Να σας υπενθυμίσω ότι ξεκινάμε την απογευματινή συνεδρίαση νωρίτερα στις 14.30.